Για uh, κόλεξ Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με το σημείο 6. Η φόρτωση των... Ε, η επιβολή τελών... Η επιβολή τελών των ε, οχημάτων των βαρέων οχημάτων ε, σε ό,τι αφορά την ε, φορολόγηση των ε, οχημάτων και την αναθεώρηση κάποιων διατάξεων. Ο κύριος Φέρμπερ είναι ο εισηγητής. Υπάρχουν τροπολογίες από την Επιτροπή Τραν. Δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, μια που έχουμε ψηφοφορία και πρέπει να περάσουμε σε αυτή το συντομότερο δυνατόν. Η πρόταση Κομισιόν αποτελείται από δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι το, η λεγόμενη Ευρωβινιέτα με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των ε, τελών κυκλοφορίας για τα βαριά οχήματα. Με τους ε, σκιώτες συζητητέ, έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε στο ότι θα σε επικεντρωθούμε στο θέμα της φορολόγησης και ε, δεν θα αντιδράσουμε στην πρόταση για την Ευρωβινιέτα, διότι δεν είναι αρμοδιότητα αυτή τη Επιτροπή. Ε, παρά τη Επιτροπή Μεταφορών, η οποία ασχολείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα με αυτό το θέμα. Και εμπιστευόμαστε λοιπόν την κρίση του. Γι' αυτό θεωρούμε πω είναι πολύ λογικότερο να επικεντρωθούμε στι κύριε αρμοδιότητε τη Επιτροπή μα, δηλαδή τη φορολόγηση. Γι' αυτό στο σχέδιο έκθεση επικεντρώθηκα σε αυτό στην ε, πρόταση δηλαδή σταδιακή κατάργηση των τελών κυκλοφορίας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, περιλαμβάνει πέντε βήματα σταδιακή κατάργησης μέχρι ε, την οριστική κατάργηση των τέλων κυκλοφορίας. Όμως αυτό θα προσθέσει διοικητικό φόρτο. Η δική μου πρόταση είναι να υπάρχει ένας ελάχιστος φορολογικός συντελεστής ο οποίος μετά από πέντε χρόνια θα μηδενιστεί. Υπάρχουν ε, πολλές τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δεν έχουν επικεντρωθεί όμως μόνο στα φορολογικά ζητήματα, αλλά καλύπτουν όλο το εύρος ε, της ε, πρότασης και μάλιστα πολλές φορές αρμοδιότητες της Επιτροπής Μεταφορών και όχι μόνο της δικής μας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να μην συμπεριληφθούν αυτές οι τροπολογίες, διότι είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Μεταφορών και προτείνουμε τη οι τροπολογίες στις δικές μας να υιοθετηθούν χωρίς ε, τροποποίηση από την Επιτροπή Μεταφορών στο σχέδιο έκθεσης. Επίσης, στην γνωμοδότηση επικεντρωνόμαστε περισσότερο στην ουδετερότητα μέχρι την ε, σταδιακή εισαγωγή της ε, Ευρωβινιέτας. Νομίζω πως ο συμβιβασμός στον οποίο έχουμε καταλήξει είναι αρκετά ισορροπημένο. Έχουμε δώσει έμφαση στις αρμοδιότητες τη επιτροπή ε, ΕΚΟΝ και χάρηκα πάρα πολύ για την καλή συνεργασία και ελπίζω σε ακόμα καλύτερη στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε. Περβάνς Μπερές. <coughs> Ευχαριστώ. Επειδή έγινε συζήτηση και με άλλους και συμμετείχα, γι' αυτό βρέθηκε κάποιος συμβιβασμός. Η βασική δυσκολία που έχουμε με αυτό το θέμα και το τομέα είναι αυτό που προτείνει να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνει 20% σταδιακή και πολύ αυστηρή κατάργηση ανά έτος. Το σημείο αφετηρίας όμως στα διάφορα κράτη-μέλη δεν είναι το ίδιο. Υπάρχουν χώρες που έχουν ήδη διόδια και τέτοια συστήματα, ενώ άλλα δεν έχουν. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που ετοιμάζονται τώρα να τα εγκαταστήσουν. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε την αρχή της ελαστικότητας που να επιτρέπει στα κρατη να διοργανωθούν προς το phasing in ή το phasing out, τη σταδιακή ε, εισαγωγή ή μείωση για τη φορολόγηση των οχημάτων των ε, βαρέων φορτηγών. Ε, υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία πρώτα απ' όλα. Υποχρέωση διέλευση, μάλλον περάσματο στο εναλλακτικό σύστημα που συζητιέται στην ΤΡΑΝ από το 2024 και ο ρυθμός μείωσης του υπάρχοντος συστήματος φορολόγησης που θα πρέπει να ε, προσαρμοστεί στο κατά πόσο προχωρά ε, το εναλλακτικό σύστημα και κατά πόσο καλλιεργείται και αναπτύσσεται, για να μην υπάρχει απώλεια εσόδων για τα κρατη Και στην ομάδα μας θα ψηφίσουμε και την τροπολογία 22 της κυρία Κοτκάτο, μια πολύ χρήσιμη τροπολογία, που είναι κατά κάποιο τρόπο ένα εργαλείο για τον προπολογισμό. για να μην συνεχίσουμε να έχουμε οχήματα ντίζελ. Ευχαριστούμε για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ο κύριος Τρεμόζα. Uh, Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει να περάσουμε στις ψηφοφορίε, υποστηρίζουμε την γενική ιδέα να περάσουμε από τα ετήσια τέλη σε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται ε, στην απόσταση που διανύεται. Πιστεύω ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό και από οικονομική και από ενεργειακή σκοπιά. Αλλά δεν συμφωνούμε με το συμβιβασμό ε, διότι ε, δεν συμφωνούμε για τα λεγόμενα ε, διόδια που θα γίνουν σε κάποια κράτη. Ποιο θα τα πληρώσει αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις Σκοτ Κέιτο. Η κυρία Σκοτ Κάτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η θέση μας για το θέμα αυτό είναι γνωστή. Θα πολύ σύντομα να την επαναλάβω. Η θέση μας είναι ότι δεν στηρίζουμε την έκθεση αυτή. Ούτε τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτού. Δεν θεωρούμε ότι θα ήταν επικοδομητικό να καταργήσουμε την ετήσια προλόγηση των οχημάτων από την ομάδα μας. Πιστεύουμε ότι τα τέλη αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιβληθούν τέλη ανάλογα με την ε, απόσταση. Πώς διανύεται και ότι πρέπει να επιζητήσουμε ε, καθαρότερες λύσεις, οικολογικότερες και για να μειώσουμε το κυκλοφορικό. Αυτά τα τέλη που βασίζονται στην απόσταση είναι ε, χρήσιμα για κάποιες περίπτωσεις περιβαλλοντικών σκοπών, αλλά δεν πιστεύουμε ότι συνολικά για τον κύκλο ζωής των οχημάτων, για περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους μπορεί να είναι χρήσιμα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα βρούμε μια βιώσιμη λύση, συμπεριλαμβάνοντα την αντιμετώπιση του αντικτύπου του κύκλου ζωής των οχημάτων στην οικονομία, τις κοινωνικές πτυχές αυτής και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρέπει επίση να δούμε το πώ αυτό σχετίζεται και με τι κλιματικέ αλλαγέ και τη χρήση άλλων εγκαταστάσεων όπω την περίπτωση των εταιρικών οχημάτων. Έχουμε λοιπόν υποβάλει τροπολογίε για να αλλάξουν κάποια πράγματα στο παράρτημα και να μην αλλάξει ο φορολογικό εντελεστή ε, σε μηδέν το 2024 όπω προτείνει ο συγητή. Ευχαριστούμε κυρία Λόπε Μπερμέχο. No opinion. E Δεν θέλει το λόγο το e INF. Floor back to rapporteur. Ο λόγος πίσω στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει γενικότερη συμφωνία απόψεων. Ελπίζω όμως ε, να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση την οποία θα μεταφέρουμε στην Επιτροπή Μεταφορών. Η πολιτική μεταφορών και η Ευρωβινιέτα δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μέσα την Επιτροπή μας. Υπάρχει ένα ε, σχετικό ψήφισμα το οποίο προετοιμάζουμε για την ε, πρόταση της Επιτροπής γι' αυτό, για την Ευρωβινιέτα και θα κλείσω λέγοντας ότι συστήνω να επικεντρωθούμε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγινε και μια συζήτηση για το κατά πόσο είναι παραδεκτές κάποιες τροπολογίες. Ε, συγγνώμη, γι' αυτό αφαιρέθηκα και δεν παρακολουθούσα. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Διακοπή ενός λεπτού. then Επειδή ελέγχουμε ένα νομικό ζήτημα για την πρώτη έκθεση, θα αρχίσουμε να ψηφίσουμε τις υπόλοιπες ε, και όταν θα μας δώσουν την απάντηση θα ψηφίσουμε την, την άλλη στο τέλος. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Ένας τελευταίος. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Και ξεκινάμε τώρα. Θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Βιέγκας ε, για μία απόφαση του Συμβουλίου για συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας. Ψηφίζουμε ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας επιπλέον από το ΕΛΚ. Ωραία. Πέρασε της ψηφοφορίας. 49 υπέρ, ένας κατά μία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα Περνάμε στην ε, έκθεση της Μόλις Κοτκάτο Κάτω για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Συμβαστική τροπολογία α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ, κατά, επαλήθευση για την 74, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για την 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. συμβασική τροπολογία Β με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίζετε λίγο γρήγορα, σας περιμένουμε μεν, αλλά τελειώνεται. Ωραία λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται συμβαστική τώρα τροπολογία χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Αν θέλετε μπορούμε να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση, νομίζω ότι απορρίπτεται. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 94 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, ήσασταν όλοι υπέρ. Λάθος δικός μου. Εγκρίνεται. Νόμιζα ότι το ΕΛΚ ήταν κατά. Ε, πρέπει να σας εμπιστεύομαι περισσότερο. Συμβαστική τροπολογία C, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 106, υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία D, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 118, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία E με προφορική τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται η προφορική τροπολογία, επομένως ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία E Θέλετε παλήθευση. Ε, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την προφορική τροπολογία. Θα δείτε όμως. πέρες ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία χωρί την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία F, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία H, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 174 με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 175, α, ψηφίζουμε την 175 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία I, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τοπολογία J, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ. 204 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για τη 204. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία και υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά α, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 211 υπέρ, κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε να το παληθεύσουμε. Πέρας ψηφοφορίας, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 213 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε παλήθευση? Όχι. Συμβαστική τροπολογία L υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία M υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 228 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία N με προφορική τροπολογία. Με την προφορική τροπολογία λοιπόν υπέρ, κατά, επαλήθευση, άρχεται ψηφοφορία. πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Επομένω ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο υπέρ. Το ΕΛΚ υπέρ φαντάζομαι. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 241 σε διάφορα τμήματα. σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, επαλήθευση, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, που είναι το 2-2 στην ουσία, επειδή απορρίπτεται, όλα τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Επομένως, περνάμε στη 2.42. Υπέρ, κατά, ποχές, εγκρίνεται. 2.43. Υπέρ, κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται να το επαληθεύσουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η 244 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία O με προφορική τροπολογία. Είπα A, συγγνώμη. O λοιπόν. Λάθος το πρόφερα. Με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Επαλήθευση της ψηφοφορία. Ένας επιπλέον από το ΕΛΚ. τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία O, λοιπόν, χωρίς προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Π, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 264, υπέρ, κατά, επαλήθευση, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της Εγκρίνεται. 265 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ. Κατά. Επαλήτευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Q υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 278 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ, κατά επαλήθευση για τη 279. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 280 υπέρ, κατά Επαλήθευση για τη 280, έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία R, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 292 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 293 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 294 υπέρ κατά επαλήθευση για τη 294 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 295 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 297 υπέρ κατά αποχές η Γκου είναι κατά, επομένως απορρίπτεται 200 να το επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται η 2.97 ήταν αυτή, έτσι. Α, συγγνώμη, η 2.96. Η 2.97 ήτανε τη τροπολογία της μόλις κάτω. Εγώ 57. Θέλετε επαναλάβουμε τη 297. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεν αλλάζει το αποτέλεσμα, απορρίπτεται ούτως ή άλλως. 2,98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2,99 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 300 υπέρ. Κατά αποχέ επαλήθευση. Άρχεται η αλλω 298 υπερ κατα αποχες εγκρινεται Πέρας ψηφοφορίας. η ψηφοφορια περας ψηφοφορία. απορριπτεται Συμβαστική τροπολογία S υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 311 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 312 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 314 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 315 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 20, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο ε, αιτιολογική έκθεση 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική έκθεση 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 5 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Δεν ξέρω αν θέλετε να επαληθεύσουμε. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Αρχικό κείμενο αιτιολογική έκθεση 5. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ο, τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ κατά αποχές, η φιλελεύθερη είναι υπέρ, εγκρίνεται λοιπόν, τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 10 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά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 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά. Δεν βλέπω τις ομάδες. Άρχεται η ψηφοφορία για την μετεωρολογική έκθεση 20, αρχικό κείμενο. Πολλές μετεωρολογικές εκθέσεις έχουμε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο ε, πλειοψηφία. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 15 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 26 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει συγγνώμη, πρέπει να πάω στο 18, τροπολογία 18 και 40 και 20 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 30 Τροπολογία 19 υπέρ κατά επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. Τη λογική αναφορά 31 υπέρ κατά επαλήθευση. Δεν βλέπω τα χέρια σας. 31 υπέρ. Ναι, άρχεται η ψηφοφορία, συγγνώμη. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 γιατί άλλες καταπίπτουν, υπέρ, κατά, επαλήθευση για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά, 26 είναι ταυτόσημη, 27, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 27. Ποπτεύομαι ότι δεν είναι δυνατόν γιατί έχω διαφοροποίηση. Το S&D είναι όλοι υπέρ αλλά οι άλλες όχι. Οι 27 υπέρ αποχές 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 36 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική αναφορά 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική τροπολογία T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 53 υπέρ κατά Επαλήθευση για την 53, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, επαλήθευση για την 56, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, Επαλήθευση για το 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το κείμενο, στροποποιήθηκε, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 42 υπέρ, 9 κατά, 3 αποχές, συγχαρητήριο στον εισαγητή. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση του Μαρκού Φέρμπερ για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Συμβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά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 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές έλεγχος έλεγχος για την 22 άρχεται ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται με, μεγάλη, με μικρή πλειοψηφία. 23 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται. Πρόταση τη Επιτροπή όπω τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία έρχεται αυτή. Πέρας. 36 ε, υπέρ, 15 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια. Έχουμε ακόμη μια ψηφοφορία. Συγχαρητήρια. Δύο λεπτά διακοπή πριν την τελευταία ψηφοφορία. Πρέπει μισό λεπτό να μιλήσω με την νομική υπηρεσία για διατροπολογίες. Δώστε μου ένα ή δύο λεπτά. in Έτσι κι αλλιώς είμαστε μπροστά σε σχέση με το πρόγραμμα. Προχωρούμε. Πάμε στην έκθεση Μπάλτς Μπερές. Καθορισμός της έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Είστε έτοιμοι. Ωραία. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Ετελογικές αναφορές 1α, αύκο 3 και 4 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Budget 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 των συνεισηγητών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 καταπίπτει. Budget 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Ναι, ναι, είναι ονομαστική. Ως συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Πέρας. 53 υπέρ, μία ψήφος κατά, 0 αποχές. Και τώρα το νομοθετικό ψήφισμα. Παράγραφος 2 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 κατά, κατέπεσε. 10 την ψηφίζουμε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο για το ίδιο δάφιο κατέπεσε. Αρχικό κείμενο 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, πρέπει να ψηφίσουμε. Ναι, ναι, σωστά. Ναι, γιατί απορρίφθηκαν όλε. Ναι, ναι, μπερδεύτηκα. Ότι η εννέα καταπίπτοντα συμπαρέσυρε την άλλη. Αρχικό κείμενο, παράγραφο 5. Υπέρ κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Παράγραφο 6. Υπέρ κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο θα το ψηφίσουμε. Ωραία, το ψηφίζουμε. Με παράγραφο 7 αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αύκο 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 και 18 καταπίπτουν. Αρχικό κείμενο και πάλι για το, 18, το τροπολογία 18 υπερκατά αποχές απορρίπτεται. Άρχικο κείμενο υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπερκατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα θεωρείται εγκριθέν όπω τροποποιήθηκε τώρα. Ε, την εντολή για να περάσουμε σε διαθεσμικές διαπραγματεύσεις με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται αυτή. Πέρας. 52 πέρα ένας κατά, μία αποχή. Η έκθεση και η απόφαση εγκρίνεται συγχαρητήρια και για τα δύο στους συνεισηγητές. Τώρα ολοκληρώσαμε. Θα επιστρέψουμε στις τέσσερις και μισή ακούγεται. Α, όχι, όχι, δυόμιση. Yeah. Ah, because it is not in the agenda. Okay, sorry. We Δυόμιση έχουμε τη δημόσια ακρόαση. Oh, uh, Και στη μία έχουμε την ομάδα εργασίας. Ευχαριστώ πέρασε.